Ladies and gentlemen, good morning everybody. As I could see... Καλημέρα σε όλους. Ε, δεν βλέπω πάρα πολλά μέλη της Επιτροπής μας ε, για να παραστούν ήδη στην αρχή της ακρόσης. Είμαι σίγουρος ότι σε 3-4 λεπτά θα προσέλθουν. Καλώς ορίσατε. Ε, κύριε Μοέντας, επί... κατόπιν απόφασης ε, του κυρίου Ζαν Κλοντ Γιούγκερ θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο ε, της έρευνας ε, επιστήμης και καινοτομίας. Η πολιτική έρευνα ε, και καινοτομία καλύπτει την έρευνα και την τεχνολογία καθώς και την διάδοση και αξιοποίηση των πορισμάτων ε, ε, των ερευνών. Οι προτεραιότητες μας συμπίπτουν απολύτως με το πρόγραμμα ε, του Επιτρόπου για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είμαστε η μοναδική επιτροπή που διοργανώνει την ακρόαση. Θα τα καταφέρουμε, δεν ανησυχώ. Ίσως ε, να παραστούν και κάποιοι συνάδελφοι από άλλες επιτροπές. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της ε, Κοινωνίας των Πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους δημοσιογράφους, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκπροσώπους ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που ασχολούνται με την έρευνα και όλους όσους παρακολουθούν τη σημερινή ακρόαση αναμεταδίδεται ζωντανά εξάλλου και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω όλους τους ακροατές λοιπόν. Ε, στρατηγική εξόδου από την κρίση. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα και με ο μεγαλύτερος, ε, η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη είναι η έρευνα. Για πολλά χρόνια προσπαθήσαμε να προωθήσουμε την έρευνα, διότι ασχολούμαστε εδώ στην Επιτροπή μας με το μεγαλύτερο στον κόσμο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, αριθμό 8 σήμερα, που φέρει τον τίτλο Ορίζοντας 2020. Είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, ε, πρόγραμμα καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ε, επίσης, μας απασχολεί πάγια το ζήτημα των νέων τεχνολογιών. Προωθούμε το λεγόμενο τρίγωνο της γνώσης. Ε, γνώση, καινοτομία και παιδεία. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της ακρόασής μας. Το πώς θα ενεργήσει την επόμενη πενταετία ο κύριος Μοέδας αν αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο αφού πρώτα σας υπενθυμίσω ε, τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα 16 για την ε, ε, διεξαγωγή των ακροάσεων. Δύο είναι βασικές ερωτήσεις. Ε, ε, έχετε την επαγγελματική επάρκεια για να μετάσχετε στο συλλογικό σώμα τη Επιτροπής και έχετε επάρκεια για να επιτελέσετε ικανοποιητικά τα καθήκοντα που θα σας ανατεθούν. Αυτά είναι τα δύο βασικά ερωτήματα. Ο υποψήφιος επίτροπος απήντησε γραπτός σε αυτά τα προπαρασκευαστικά ερωτήματα Πέντε είναι συνολικά και τα δύο είναι ίδια για όλες τις επιτροπές. Ε, τρία σχετίζονται με τα, τα θέματα αρμοδιότητας της επιτροπής μας. Τα έχετε λάβει, υπάρχουν και στην ιστοσελίδα. Επίσης έχετε ε, το βιογραφικό σημείωμα, ε, την επιστολή για την αποστολή του, τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, καθώς και την επιστολή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που πιστοποιεί ότι η δήλωση οικονομικών συμφερόντων του κυρίου Μουέντας εξετάστηκε και εγκρίθηκε. Και έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Πώς θα διεξαχθεί η ακρόαση. 15 λεπτά για την αρχική εισαγωγική παρουσίαση του Επιτρόπου και στη συνέχεια ε, τελική παρουσίαση κατόπιν ε, πεντάλεπτες ερωτήσεις ε, από πλευρός των βουλευτών βάσει της αρχής του πινκ πονγκ. Ερώτηση, απάντηση, ερώτηση, απάντηση. τρία λεπτά για ερώτηση, δύο για απάντηση. Ο πρώτος γύρος από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και σας ενημερώνω ότι ε, παρέχετε διερμηνία σε 23 γλώσσες, 23 πέσιμε γλώσσες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη μητρική σας εκ τούτου. Παρακαλώ να τηρήσετε το χρόνο αγόρευσης όπως θες. Θα μαγνητοφωνηθεί και η ακρόαση. Στην ίδια ιστοσελίδα θα είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να ακούσετε και τις χθεσινές ακροάσεις ήδη. Θα αρχίσουμε τώρα. Θα δώσω το λόγο στον υποψήφιο επίτροπο για 15 λεπτά. Παρακαλώ.